Τώρα, περνάμε στις ε, δηλώσεις ψήφου. Επεξηγής ψήφου, με συγχωρείτε, επεξηγής ψήφου. Και δίνω το λόγο στον κύριο Άλντο για ένα λεπτό. Presidente, L'onorevole Patriciello. Sì, Presidente. Prego, chiedo ai colleghi di lasciare l'emiciclo per chi la vuole lasciare e consentire all'onorevole Patriciello. Λοιπόν, παρακαλώ, όσοι θέλετε να μιλήσετε, παρακαλώ να βγείτε έξω από την αίθουσα και να επιτρέψετε στον κύριο Πατριτσέλο να προχωρήσει στην επεξήγηση που θα δώσει για την ψήφο του. Ας περιμένουμε λιγάκι. Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ε, συγχαίρω τον εισηγητή ε, και όλους τους συναδέλφους ε, που δούλεψαν για να υπάρξει αυτό το νέο εργαλείο. Ένα νέο εργαλείο το οποίο θα επιτρέψει την χορήγηση μικροκονδυλίων και μικροχρηματοδοτήσεων σε άτομα και εταιρείε που έκαναν σωστά τη δουλειά τους τα τελευταία χρόνια. Ε, έχουν χαθεί 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τράπεζες ε, δεν δίνουν εύκολα δάνεια. Ως εκ τούτου το εργαλείο αυτό θα επιτρέψει σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση να την ξεκινήσουν με μεγαλύτερη ευκολία στην πρόσβαση στα απαραίτητα κονδύλια. Αυτή λοιπόν η νέα πρωτοβουλία θα συμβάλλει στο να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας οι οποίες ε, θα συνοδευτούν και με άλλα μέτρα και με άλλα κονδύλια με την κατάρτιση που θα επιτρέψει στους νέους να έχουν κάποια βοήθεια ε, σε, αυτό, τα αυτά τα ε, προγράμματα. Αυτό λοιπόν το εργαλείο κύριε Πρόεδρε πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να δοθεί μια νέα όθηση στις μικρομεσαίες εκείνες επιχειρήσεις που είναι ο παλμός ε, και η σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Στόγιανοφ Δημήταρ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι υπερψήφισα την έκθεση αυτή, γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση, πολύ κατάλληλη για τη σημερινή στιγμή και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε με μέτρα σημαντικά που υιοθετούνται και σε άλλε χώρε όπω τη χώρα μου παραδείγματο χάρη. Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πάρα πολύ ρητικό περιβάλλον για τι επιχειρήσει εκείνων που έχουν πολύ μικρέ επιχειρήσει, διότι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιστώσει από τι τράπεζε. Αυτό δεν είναι συμβατό με την ιδέα μια τράπεζα. Έχω την εντύπωση ότι οι τράπεζες εφευρίσκουν διάφορε δικαιολογίε για να μην χορηγούν πιστώσει. και εάν χωρηθούν οι πιστώσεις αυτές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να δώσουν εγγυήσεις πολύ υψηλών ε, αξιών. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα για μικροπιστώσεις και ελπίζω ότι αυτό το μεθοτικό κείμενο θα βοηθήσει την οικονομία της Βουλγαρίας συγκεκριμένα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Στότ. Uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να είναι σαφές ότι έχω την εντύπωση μεν ότι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις είναι καλή ιδέα και θα πρέπει να συνεχιστεί θα πρέπει να συγχυθεί σε εθνικό επίπεδο. Ανησυχώ λιγάκι με την πρόταση αυτή. Δεν ξέρω πώ θα αιτιολογηθούν τα χρήματα αυτά, από πού θα προέρθουν και πώ θα επιστραφούν. Θα ήθελα να ενθαρρύνω, ενθαρρύνω συγγνώμη, τις εθνικές κυβερνήσει να κάνουν ό,τι μπορούν για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, που είναι ο ακρογωνιαίο λίθος τη οικονομία μα. Και θα πρέπει οι πόροι αυτοί να διαθέτουν τίθενται σε εθνικό επίπεδο. Θα σας ευχαριστώ κύριε Τότ. Ο επόμενο ομιλητής παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε την δυνατότητα να σα εξηγήσω πώ ψήφισα. Εμεί ήμασταν υπέρ τη πρόταση αυτή, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε επιχειρηματίε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, να του βοηθήσουμε να δημιουργήσουν πλούτο και θέσει απασχόληση και να καταπολεμήσουν τη φτώχεια. Επίση χαίρομαι που ε, θα προέρχονται τα κονδύλια αυτά από το σημερινό προπολογισμό και δεν θα ζητήσουν συμβατικά κονδύλια. Θα ήθελα όμω να τονίσω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τα χρήματα του φορολογούμενου γιατί δεν πρέπει να ξέρω, ξεχνάμε ότι υπάρχουν παραδείγματο χάνει και διάφορε ενώσει στην Καραϊβική που βοηθούν τι κοινότητε, οι οποίε όμω έχουν, ε, των οποίων μάλλον τι αρμοδιότητε έχουν σφιτεριστεί οι τοπικέ αυτοδιοίκησει. Και δεν υπάρχει έτσι επαρκή πρόσβαση στι ε, μικροπιστώσει. Θα πρέπει να μην κάνουμε εμεί κάτι παρόμοιο. Ευχαριστώ κύριε Καμάλη, ο πρόεδρο. Ο κύριο Αλφρέτο Πανέλο έχει το λόγο. Ε... Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι μας ε, συμφωνούμε όσον αφορά το πρόβλημα των ε, μικροπιστώσεων. Και γι' αυτό λοιπόν όταν ε, μιλάμε για τέτοιου είδου θέματα θεωρώ ότι είμαστε δεσμευμένοι να διατηρήσουμε αυτές τις μικροπιστώσεις και να γνωρίζουμε ότι δεν οφείλουμε ότι δεν πρέπει να επεκταθεί αυτό το μέτρο και σε άλλους τομείς γιατί οι μικροπιστώσεις ε, προέκυψαν για να βοηθηθούν ε, οι λιγότερο ευνοημένοι. Ως εκ τούτου μιλάμε και για ένα πρόβλημα που έχει σχέση με τον πολιτισμό. Σε πάρα πολλές χώρες και νομίζω περισσότερο στις χώρες που το χρειάζονται, δυστυχώς δεν υπάρχει η σωστή πολιτιστική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να αποκτήσουν αυτές τις πιστώσεις. Εγώ λοιπόν είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι αυτά τα εργαλεία θα πρέπει πρώτα να ε, αποκτηθούν από τις κυβερνήσεις που τα χρειάζονται. Υπάρχουν στην Ευρώπη δύο ταχύτητες. Αυτές ε, οι χώρες που είναι η Γερμανία και η Γαλλία και η δεύτερη ταχύτητα είναι οι χώρες εκείνες που έπρεπε να έχουν διαφορετική πολιτιστική προσέγγιση στο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που διακυβεύεται, το πραγματικό πρόβλημα στην Ευρώπη ε, δεν είναι ότι υπάρχει μόνο το θέμα της χρηματοδότησης, ότι είναι δύσκολη η χρηματοδότηση. Ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οφείλουμε να ε, δώσουμε τη δυνατότητα να εργάζονται κυρίως αυτοί που όπως σας είπα είναι οι λιγότεροι ευνοημένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουν ζητήσει άλλη το λόγο για επεξηγήσεις ψήφου. Ε, διακόπτουμε, θα ξανασυνεχίσουμε στις 3. Γεια σας και καλή σας όρεξη, εύχεται ο Πρόεδρος.